Θα προχωρήσουμε τώρα στις ε, επεξηγήσεις ψήφου. Καλό όλους τους βουλευτές ε, που θέλουν να φύγουν από την αίθουσα και που δεν ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη συζήτηση να φύγουν ησύχως. Σας ενημερώνω ότι έχω λάβει διάφορα αιτήματα για επεξηγήσεις ψήφου και μπορούμε να συνεχίσουμε όμως μόνο μέχρι τις 14.45 το αργότερο για να μπορέσουν οι υπηρεσίες να προετοιμάσουν την επανάληψη της συνεδρίασης στις 3. Όλες λοιπόν οι αιτήσει για αιτιολόγηση ψήφου θα, θα εξεταστούν ε, και οι υπόλοιπε θα υποβληθούν γραπτός όσες δεν μπορέσουν να γίνουν προφορικός. Ξεκινάμε την έκθεση Μόησα. Ησυχία παρακαλώ. Αναλαμβάνει στα γαλλικά ο Πρόεδρος όσοι δεν ενδιαφέρονται για τη συζήτηση παρακαλούνται να αποχωρήσουν. Πότσακ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι πεπισμένος ότι δεν θα γίνει ακουστή η φωνή μου, αλλά παρόλα αυτά θα μιλήσω. Χαίρομαι για την προσέγγιση που έχει επιτευχθεί με τη Μολδαβία από την εποχή που ήμουν ήδη μέλος